Συνάδελφοι, είναι η ώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες και αρχίζουμε με την πρώτη έκθεση στον κατάλογο ψηφοφοριών που είναι το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη η έκθεση της κυρίας Γκαρντίνη για σύναψη τροποποίηση τη Δόχα στο πρωτόκολλο του Κιώτο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή κλπ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε έναν παραπάνω του FDD, του EFDD. Okay. Il voto è Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια την κυρία Γκαρντίνη. Πάμε στο επόμενο σημείο. Έκθεση Λαβία όσον αφορά την πρόταση του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας με την Ισλανδία. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι που ξεκινάει τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνατε λοιπόν. Eh, Πάμε στην έκθεση συναδέλφου Γκριζή όσον αφορά το περιορισμό των εκπομπών ορισμένων μέσων στην ατμόσφαιρα. Πάμε στη συμβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. It is quite clear. But if you want... Είναι σαφές. Αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε αυτό που θέλετε. Καλώς. Και τώρα πάμε συμβαστική 1. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχους. Έχουμε έναν ΕΛΚ παραπάνω. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα τη συμβιβαστική 2α. Δύο α υπέρ, δύο α συμβαστική κατά, έλεγχος. Έχουμε έναν S&D παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 2β. Υπέρ, κατά, αποχές, ας κάνουμε έναν έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 137, 22 και 17 της Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία, ο ηλεκτρονικό έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε έναν ΕΛΚ παραπάνω. Ένα μέλο του ΕΛΚ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. μαζί 23, 11, 139, 199, 218, 247, 263. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 150 ριβαζή έκια και φορέντσα. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ένας ΕΛΚ παραπάνω. Πέρας. Απορρίπτεται. «162» υπέρ της τροπολογίας «162» κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την 179 σαν προστίκη στη συμβαστική 10 Ριβασί, Πεντιτσίνι, Εκ και Φορένσα. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. Την 190, τροπολογία 190. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε την 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 196 και 197 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα Πρέπει να ψηφίσουμε την 238 πέτικα είναι. 238 υπέρ κατά απορρίπτεται. Μετά συμβιβαστική 5 υπέρ της 5 της συμβαστικής κατά αποχές εγκρίνεται. Συ, συμβαστική 7 τώρα. Υπέρ της συμβαστικής επτά. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 280. 280. Ριβασί πεντιτσίνι Εκ Φορέντσα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έχουμε έναν ΕΛΚ περισσότερο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 283 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται νομίζω αλλά σε ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πάντα έναν ελκ παραπάνω έχουμε πέρας απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 287 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 289 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. αποχές Τροπολογία 295, 296, ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 281 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 294 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 239-282 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται. Τροπολογία 292 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 160 α συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 160 υπέρ υπέρ είσαστε ελκ υπέρ υπέρ λοιπόν κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 18 υπέρ της συμβιβαστικής 18 κατά αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Έλεγχος λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 303 υπέρ 303 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 305 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, λοιπόν καταπίπτει, ψηφίζουμε τις τροπολογίες 306 και 23 ήτρε. Είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 341 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 343. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 344. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 342. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 346 και 163. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 347 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 348 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 349 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 350 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. καταπίπτουν διάφορους. Πάμε στην 370 κονέτσνα μαζί με την 372 μαζί υπέρ κατά αποχές έλεγχος περίεργες ψηφοφορίες ψηφίσατε όλοι πέρας Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 375 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 381 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 382 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 383 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ τη συμβαστική 3 κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική 6 υπέρ τη συμβιβαστικής 6 κατά αποχές εγκρίνεται. Σε αιτιολογικές σκέψεις πάμε. Ξεκινάμε από την τροπολογία 49. Παολούτσι, Καπούτο και άλλων. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 64 Δαντέν Γκροστέτ, και κλπ. Υπέρ μαζί με την τροπολογία 3 του εισηγητού και τροπολογία 3 ήτρε. Μαζί αυτές. Υπέρ. κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω. Πέρας. Εγκρίνονται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 68. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 69, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 70, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 71, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τότε τροπολογία 73, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 του συγητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα Διαλεκτρονική ψηφοφορίας ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα έκθεση. Ψηφίσατε όλοι. Ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την απόφαση για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων βάσει της εκθέσεως που ετροποποιήθη και με τη διαπραγματευτική ομάδα που απαρτίζεται από τους προέδρους και τους εισηγητές και τους κοιόδους εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων. Άρχεται η ψηφοφορία. Il voto è chiuso, avete Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Στον εισηγητή. Ε, Adesso, colleghi, passiamo Περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας ε, διάταξης. Ψηφίζουμε την έκθεση της συναδέλφου Εύη για την πρωτοβουλία για την πράσινη οικονομία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Υπέρ της τροπολογίας 1. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω έχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4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 Ψηφίζουμε την τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή, ε, τροπολογία 29 υπέρ λάθος λέει πρόεδρος, συγγνώμη, συμβαστική 3 Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ της συμβιβαστικής 12 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 Ματζουρόνης υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι οι δύο μεγάλες ομάδες καταψήφισαν έλεγχος Avete votato tutti? C'è sempre un PPE di troppo. Πάντα υπάρχει ένα μέλο του ΕΛΚ περισσότερο. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε πάλι ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβιβαστική 10 υπέρ της συμβιβαστικής 10 κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 φαρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 117 κονέτσνα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται διελεκτρονικής ψηφοφορίας, η τελική ψηφοφορία, η οποία άρχεται. Πάντα έχουμε ένα ΕΛΚ παραπάνω, πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Ψηφίσουμε την έκθεση Πιετικάνεν όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ξεκινάμε από την τροπολογία 48 για απόρριψη της προτάσεως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία ένα μέλος του περισσότερο ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται ψηφίσουμε τώρα την 145. Υπέρ της 145 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 146 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 149 υπέρ α συγγνώμη πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 156 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, αλλά βλέπετε είναι διασκορπισμένες οι ομάδες εδώ και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Τροπολογία 166, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 167, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 172. Λάθος λέει ο πρόεδρος. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 179 υπέρ ...179 υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται... ...συμβιβαστική 3 εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία και δίνω το λόγο στην συγγήτρια. Προφορική τροπολογία διαγράφει το ακόλουθο κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε, για μια μεταβατική περίοδο 20 ετών με, με το ενδεχόμενο παράτασης. Το έχουμε διαπραγματευτεί και με τους άλλους κοιόδης εισηγητές. Καλώς υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 3 με την προφορική τροπολογία της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 192, 193, 194, 195 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 196. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 201 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 201. Ψηφίσατε όλοι. Πάντα έναν παραπάνω του έλκα έχουμε. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 14, 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 214 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 216 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ της 4. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 225 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 228 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 230 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 232 υπέρ καταπίπτει διότι απορρίψαμε τη 226. Ψηφίζουμε τη 234 υπέρ της 234 κατά αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ κατά α, αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά α, αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τώρα τη 237 υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται 238 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 240, 241 και 242 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 6 υπέρ τη συμβιβαστική 6 κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, Τροπολογία 245, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 244 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 246. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, ψηφίσαμε τη 246 που κατέπεσε. Απερίφθεια λέει είχε καταπέσει. Διότι είχαμε απορρίψει τη 245. Τώρα ψηφίζουμε την 247 και την 248 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Ψηφίζουμε. Έλεγχο θέλετε. Καλώς. Ας ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 249, 250 και 251 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 255 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 256 σόμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 257 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 258 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 259 Επέρ. κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 275. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 277. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 281. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 282. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 289 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες 296, 297 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία αυτή καταπίπτει 299 γκαρντίνι υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 18, συγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 308 Dortmund. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 313 υπέρ 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 322 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 323 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 324 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 330 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 332 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 331 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 363 του συναδέλφου Ντόρμαν. 363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 365 πάντα του συναδελφού Ντόρμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 373 Άουκεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 385 Γκαρντίνη. Υπερ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 392 του συναδέλφου Ντόρμαν. Υπερ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 393 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 396 Γκαρντίνη υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 401 Ντόρμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 402. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μαζί τώρα τις τροπολογίες 406 και 407. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 409 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 411 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 412 υπέρ κατά Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Α. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 1 τώρα. Υπέρ της συμβιβαστικής 1. Κατά. Εγκρίνεται. Ποιος απέχει. Εγκρίνεται. Έλεγχος. πέρας εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ α συγγνώμη ο πρόεδρος 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Συμβατή με μια προστίκη υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 και 79 τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, Τροπολογία 6. 6 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 109, διότι 107 και 108 και κάποιες αντίστοιχες τροπολογίες έχουν απορριφθεί. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 109 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 116 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 126 διότι όλες οι προηγούμενες καταπίπτουν τροπολογία 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ της 129 κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Τελειώσαμε. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός πώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και έχουμε την έκθεση της συναδέλφου, την συναδέλφου Πατριτσέλο. Allora, colleghi, il, eh, eh, votiamo adesso l'opinion del collega Prasid. Ψηφίζουμε τώρα τη γνωμοδότηση Πατριτσέλο όσον αφορά τις διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά τις ακροάσεις των επιτρόπων. Ψηφίζουμε παρευθύ στην τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαναλάβω. Τροπολογία 21. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 26 με μία προφορική τροπολογία από πλευρά σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η προφορική τροπολογία το ότι πάντα είναι εγγυημένε με το έχουν. Always uh, be guaranteed they have. Και τονίζει ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλήρη εξαντλητική απάντηση από τους υποψηφίους ε, επιτρόπους. Έχετε αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν αντίρρησεις. Ψηφίζουμε τροπολογία 26 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συμβαστική 2 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία 33 με, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ας γίνει έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε. Συμβιβαστική 3. Υπέρ της συμβιβαστικής 3. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το τροποποιηθέν κείμενο ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια, συνάδελφε Πατριτσέλη. Διακοπή δύο λεπτών. Ούτως ώστε εκείνοι που θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να μπορέσουν να το κάνουν και θα συνεχίσουμε. συνάδελφοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε, δηλαδή να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Είχαμε μακρά ψηφοφορία σήμερα, αλλά τελειώσαμε. Και ξαναρχίζουμε με το έργο της Επιτροπής μας εκτός από τις ψηφοφορίες. Και πάμε συγκεκριμένα στο σημείο 14 που αυτό είναι μια γνωμοδότηση προς τη νομική επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνω αμέσως για αυτό το θέμα το λόγο στην συντάκτρια γνωμοδότηση, στην κυρία Γκούτελαντ και μετά θα ακούσουμε, θα κάνουμε τον πρώτο γύρο σχολείων και γνωμών με του σκιώδη των πολιτικών ομάδων. Να χαιρε... καλωσορίσω όμως, πριν αρχίσουμε, κάποιους ε, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο. Η συνάδελφοι Αρμάου, ο συνάδελφος Αρμάου, τους κάλεσε και ήρθαν να δουν πώς εργάζεται η Επιτροπή μας. Κυρία Γκούτελαντ, έχετε το λόγο για την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι βεβαίως μια πρόκληση να αρχίζουμε αυτό το θέμα μετά από τη μακρά ψηφοφορία, όμως χαίρομαι γιατί αρκετοί συναδελφοί έμειναν. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση που θα πάει στη Νομική Επιτροπή, όπως είπε και ο Πρόεδρος, και πρόκειται για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Είναι σημαντικό ότι κάνουμε και εμείς στην Επιτροπή μας αυτή τη συζήτηση. Κάθε μέρα στο Κοινοβούλιο κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξουμε τις περιβαλλοντικές πολιτικές, να αποφασίσουμε για τις νομοθεσίες. Μετά όμως τι γίνεται. Πολλές φορές οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητούμε πολύ πιο συχνά. Μία πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές αργούν να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο της, ε, ε, τα νομοθετήματα, μετά υπάρχουν καταγγελίες που αντιμετωπίζονται από την Επιτροπή Έχουμε επίσης ε, τον έλεγχο που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά έχουμε τις διαδικασίες επί παραβάση, όπου η Κομισιόν προσφεύγει κατά των κρατών μελών στα δικαστήρια. Υπάρχει επίσης το θέμα αν είναι ε, κατάλληλη νομοθεσία. Εδώ έχουμε το REFIT. Εγώ θα εστιάσω στη νομοθεσία της Ένωσης που είναι σημαντική για τη δική μας την Επιτροπή του Περιβάλλοντος, την Ένωση. Δηλαδή η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται που έχει προτεραιότητα στο 7ο πρόγραμμα ε, δράσης. Πολλά κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν πολλές ευθύνες όταν πρόκειται για την εφαρμογή της ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία δεν εφαρμόζεται καθόλου πολλές φορές αυτή η νομοθεσία ή πλημελώς. Ε, η έκθεση της ε, Επιτροπής που συζητάμε δείχνει ότι περισσότερες περιπτώσεις ε, που απασχόλησαν την Κομισιόν για την καθυστερημένη εφαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο, 168 αφορούν το περιβάλλον, 158 το θέματα υγείας και καταναλωτών και υπήρχαν σαφή παραδείγματα καθυστερημένης ε, ε, ε, μετάθεσης μεταφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο τις οδηγίες για τις εκπομπές. Οι, οι δεύτερες συχνές καταγγελίες αφορούν το περιβάλλον. Το 2013 ο μεγαλύτερος αριθμός διαδικασιών επί παραβάση αφορούσαν το περιβάλλον και νέες διαδικασίες επί παραβάση αλλά και αιτιολογημένες γνώμες. Χίλιες ε, 334 διαδικασίε επιπαραβάση αφορούσαν το περιβάλλον. Μεγάλε οι προκλήσει λοιπόν όταν πρόκειται για την εφαρμογή τη περιβαλλοντική νομοθεσία σε επίπεδο ενώσεω. Κατά τη γνώμη μου και καλό την Επιτροπή να συνεχίσει την ε, τυπική διαδικασία επιπαραβάση, ιδιαίτερα όταν οι άτυπες συμφωνίες δεν λειτουργούν. Επίσης, το θέμα της εφαρμογής και της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δεν πρέπει να σημαίνει ότι μειώνουμε τις, φιλο... τις φιλοδοξίες μας όταν πρόκειται για την πολιτική υγείας και περιβάλλοντος. Ε, υπάρχει επίσης μεγάλος χρόνος διαχείρισης ε, για τις πολιτικές. ή οργανώσεις των πολιτών ε, θα πρέπει να, δηλαδή είναι, ε, ε, ε, δικαιούνται να αναμένουν ταχύτερη διαδικασία. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο για να ιεραρχούνται από την Κομισιόν στρατηγικές υποθέσεις μεγάλου ενδιαφέροντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί έχει πεπερασμένους πόρους, άρα πρέπει να κάνει μια στρατηγική. Τώρα, για την απλούστευση της νομοθεσίας ...το πρόγραμμα REFIT που έκανε η Κομισιόν, θέλω να υπησέλθω σε αυτό και λεπτομερώς να αναφέρω κάποιες άλλες προτάσεις. Όμως το REFIT δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει πρόσχημα για να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας στην περιβαλλοντική προστασία και την ασφάλεια των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρομαι σε αυτό που λέμε gold plating, που μεταφράζεται ως ε, κανονιστικός υπερθεματισμός, υπερβολή δηλαδή στους κανονισμούς. Πρέπει να ε, το ορίσουμε καλύτερα τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί καλό είναι να κριτικάρουμε τη βαριά νομοθεσία και τις ρυθμίσεις, αλλά από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες αν ε, είναι μόνο ελάχιστοι οι κανόνες που έχει μέχρι τώρα. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ενωσιακού και επίπεδου κρατών μελών, ούτως ώστε να είναι και η νομοθεσία ε, ισορροπημένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Βάντεν Καϊντελάιεν από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πρότασή της σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Όπως φαίνεται στην ετήσια έκθεση, κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και η χώρα μου, το Βέλγιο, σίγουρα δεν είναι από τους καλύτερους μαθητές στην ευρωπαϊκή τάξη. Η απόφαση ε, σύνταξη γνωμοδότηση για πρώτη φορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, σηματοδοτεί κάτι πολύ σημαντικό. Εμεί θα υποβάλλουμε εξ ονόματος ομάδας με τροπολογίε για να καλύψουν, θα καλύψουν τα τρία βασικά που θέλω να πω στην εισηγήτρια. Για τον έλεγχο τη εφαρμογή τη περιβαλλοντική νομοθεσία με το νέο πιλωτικό πρόγραμμα η Κομισιόν ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να παρακολουθεί περισσότερο και πιο, από πιο κοντά τη συνεργασία με τι εθνικέ περιφερειακέ τοπικέ τις αρχές. Δεύτερον, να προσπαθήσει η νομοθεσία, να, να είναι νομοθεσίες φιλικές προς τους πολίτες και τους χρήστες και οι Κομισιόν μαζί με τους πρωταγωνιστές και τους εμπλεκόμενους εδώ να ε, μπορούν να συνεργάζονται. Ε, πρέπει να είναι πιο πρακτική η νομοθεσία. Αυτό εκφράζει τις επιθυμίες όλων των πολιτών. Τρίτον, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε την περιβαλλοντική νομοθεσία. Εγώ τονίζω την αρχή της επικουρικότητας ταυτόχρονα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η οικονομική ευημερία προέρχεται από τους ε, εναρμονισμένους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. οι κανόνες των κρατών μελών των ιδίων πρέπει να παρακολουθούνται εκ του Ευχαριστώ την συγγήτρια για την πρότασή της και προσβλέπω στη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα για την ομάδα ECR ο κύριος Τόρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Το δικαίωμα ελέγχου όταν δεν εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τις ε, συνθήκες αποτελεί ακρογωνίο λίθο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Άρα συμφωνεί με την αρχή του κράτους δικαίου, του κράτους δικαίου που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το, και το ενωσιακό δικαίωμα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υποτίθεται πρέπει να ελέγχει, δεν έχει τους πόρους ε, και τα μέσα για να χειριστεί όλες τις υποθέσεις ε, πλημελούς εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα πρέπει να γίνει πραγματικά πολιτική προτεραιότητα για την Κομισιόν όμως η εποπτεία τη εφαρμογή Νομοθεσίας και αυτό σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που, στο οποίο είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εταιρείε μπορούν επίσης να αποβάλουν καταγγελίες για τη μη εφαρμογή ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά θα πρέπει και η Κομισιόν να φροντίζει να υπάρχει διαφάνεια όταν ε, κινείται διαδικασίες επί παραβάση. Πρέπει να ενημερώνει δηλαδή τους πολίτες. Και αυτό να γίνεται έγκαιρα και ορθά. Το ίδιο ισχύει για τη συνέχεια που δίνει στις καταγγελίες η Κομισιόν. Επίσης θα πρέπει να ερευνά ιδιαίτερα τις περιπτώσεις ε, που έχουν να κάνουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Να εφαρμόζονται πιο σωστά οι κανόνες. Αυτό είναι προς όφελος των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής και βέβαια θα πρέπει να τηρούνται και αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Και σε περιφερειακό επίπεδο οι πολίτες, οι οργανώσεις περιμένουν να, να υπάρχει μια αξιόπιστη δέσμη κανόνων. Και δεν θέλουν να στρέβλωση του ανταγωνισμού, αλλά αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να τα έχει υπόψη της η Κομισιόν, γιατί οι πολίτες δυσκολεύονται και υπάρχει και πρόβλημα με την αποδομή δικαιοσύνη από τα δικαστήρια πολλές φορές. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας αν υπάρχει αλλαγή κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, ε, αν υπάρξει έλλειψη συντονισμού, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Δεν μπορεί να, εφαρμοστεί, δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι διατάξει των οδηγιών, αν υπάρξουν και ανακατατάξεις στα διοικητικά όργανα κτλ. Όλε αυτέ είναι περιπτώσει κακή εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει πολλά για την σωστή εφαρμογή των οδηγιών. και την επιβολή της νομοθεσίας εν γέννη. Ιδίω όταν καθυστερούν ορισμένα κρατημέλη να εφαρμόσουν την ενωσιακή νομοθεσία. Στην προκειμένη περίπτωση θα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει τι σχετικέ πληροφορίε μέσω μια φιλική προ το χρήστη βάση δεδομένων που θα δίνει πληροφορίε για τη μη εφαρμογή των ε, νομικών πράξεων της Ένωσης από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και να πω βέβαια ότι και εγώ περιμένω να συνεργαστώ πολύ καλά με, με την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Ο πρόεδρος τώρα, η κυρία Κονέτσινα για την ΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το σημαντικό θέμα που απασχόλησε τη συντάκτρια. Καταρχήν να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα μέσο καλής ρύθμισης ε, της λειτουργίας της Ένωσης. Πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως πρόκειται και για ποσοτικό σφάλμα εδώ, δηλαδή πρόβλημα με τον αριθμό των εκδεδομένων κανονισμών και οδηγιών που καμιά φορά προκαλούν χάος στα κράτη-μέλη. Το κείμενο είναι τέτοιο σαν να μην έχει υποχρέωση η Κομισιόν να ε, παρέχει ανάδραση, ένα feedback ε, και έναν έλεγχο για την εφαρμογή. Όμως, μέχρι τώρα ε, αναφερόταν ότι τα κράτη-μέλη έκαναν λάθος. Αυτό δεν το πιστεύω εγώ. Πρέπει να πούμε ότι και η Κομισιόν κάνει λάθη. Και αν θέλει να έχει καλύτερη εφαρμογή του δικαίου, πρέπει να κάνει και εκείνη καλύτερα τη δουλειά της. Πολλές φορές υπάρχουν αμφιβολίες και διχογνωμίες ε, στην ερμηνεία των οδηγιών. Εγώ ήμουν 12 ε, χρόνια εθνική βουλευτής και πρέπει να πω ότι αυτά που έφταναν σε εμά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν τόσο ασαφή ε, και χαοτικά που δεν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. βέβαια, παρόλο που θέλαμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή. Δεν είχαμε όμως βάση σαφή για να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις κι εμείς πολλές φορές ε, η Κομισιόν χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στις διάφορες χώρες. Αυτό που είναι αποδεκτό σε μια, από μια χώρα δεν είναι από μια άλλη. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ παλιών και καινούριων κρατών μελών, μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών μελών και η Κομισιόν τα αντιμετωπίζει διαφορετικά και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του δικαίου. Ε, σε αυτό το σημαντικό κείμενο και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και να το προσθέσουμε και να, και να πούμε ότι η Κομισιόν ε, υπερβολικά χρησιμοποιεί την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολική σε αυτό το θέμα. Καμιά φορά αυτό οδηγεί σε καταχρήσεις σε βάρος των μικρών και νέων κρατών μελών που απειλούνται σε σχέση με τα κονδύλια των ταμείων. Ακόμα και αν θα κέρδιζαν μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πολλά κράτη-μέλη ε, δεν τολμούν να το κάνουν. Και πολλές φορές δέχονται την ερμηνεία των υπαλλήλων της Κομισιόν χωρίς να ε, προσφεύγουν σε αυτή τη δυνατότητα του δικαστηρίου, γιατί φοβούνται ότι μετά δεν θα τους δίνουν καθόλου τίποτε από τα ταμεία. Επίσης η Κομισιόν ε, τους κανονισμούς και τις οδηγίες και τα άρθρα των οδηγιών ε, θα πρέπει να τα εξετάζει πιο προσεκτικά όταν εφαρμόζουν άλλα κράτη-μέλη και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή την καθαρή ατμόσφαιρα. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο μία χώρα, αλλά περισσότερες. Και αν υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή σε ένα κράτος μέλος, πρόβλημα εφαρμογής της οδηγίας, τότε ε, υποφέρουν οι πολίτες ενός γειτονικού κράτους μέλους. επειδή δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Πάλι υπάρχει ένα θέμα μικρών και μεγάλων ε, κρατών μελών. Αλλά αν η, μια, η εφαρμογή μιας οδηγίας δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία ε, πολιτών άλλων χωρών, αυτό πρέπει να το δει κατά προτεραιότητα η Κομισιόν. Δεν το βλέπω να το κάνει. Εγώ θα καταθέσω κάποιες σχετικές τροπολογίες. Δεν ισχυρίζομαι ότι ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά στηριγμένοι στη λογική. Και δεν πρέπει ε, ε υπερβολικά εύκολα να κατηγορούμε κράτη-μέλη. Γιατί πολλές φορές ε, κάποιες γενικές διευθύνσεις συμπεριφέρονται σε ορισμένα κράτη-μέλη με τρόπο απαράδεκτο. Δεν θα συνεχίσουμε να το δεχόμαστε αυτό. Σας ευχαριστώ για την ομάδα EFTD τώρα, ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν σαφώ και διαφανώ και εγκαίρω και μέσω του διαδικτύου δυνατών όχι μόνο ότι υπάρχουν νόμοι και προδιαγραφέ, αλλά και ποιε εθνικέ νομοθεσίε έχουν υιοθετηθεί και έχουν σωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Και ποιο έχει την ευθύνη να επικαιροποιήσει σωστά τις, ε, την νομοθεσία. Ο μηχανισμό του EU Pilot πάει πολύ καλά αλλά μετά σε δικασίες κατά παράβαση οι, οι, πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κατωμέλος. Έχουμε επιλοτικές υποθέσεις όπου οι επιτροπές των πολιτών που εκπροσωπούν τοπικά συμφέροντα ζητούν χωρίς επιτυχία να δουν επίας βάσος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει τις παρατηρήσεις και τι επικρίσεις. Θέλουν να δούνε πώς τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται ποτέ, όμως δεν επήραν σαφεί απαντήσει. Και τέλο, αν τα κράτη-μέλη δεν ε, ανταποκρίνονται, συμμορφώνονται. Τι ακριβώς συμβαίνει. Κατά μας είναι παράδοξο το τέλος μιας ε, δικασίας κατά παράβαση να είναι ένα πρόστιμο ε, που πληρώνει το κράτος και τελικά οι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Πληρώνουν πάντα οι πολίτες και από πλευράς υγείας πληρώνουν να μην υπάρχουν παραβάσεις που αφορούν το περιβάλλον και από ρήπανση και πληρώνουν και τη ρήπανση και μετά πληρώνουν και όταν το κάτω μέλο ε, πρέπει να υποστεί τη διαδικασία κατά παράβαση και να πληρώσει ε, ε, κάποια ποινή. Το σύστημα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει. Ποιο είναι εδώ? Ο κύριος Μπανκέμπης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που βάλατε το θέμα στη μερίσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι η πρώτη φορά και εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντό σα, διότι η εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία που πράγματι αποτελεί ψηλή λοιπόν προτεραιότητα. Και είναι μάλιστα και σε ε, περίοπτη θέση στο κατάλογο των νομοθεμάτων που δεν εφαρμόζονται. Παρθμόν 1, παρθμόν 2 για σειρά ετών και ήδη και στην ετήσια έκθεση του 2014 ε, τα πράγματα δεν θα έχουν αλλάξει. Σύντομα θα λάβετε αυτή την έκθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο καλύτερη νομοθεσία, better regulation, περιλαμβάνεται αυτή η προτεραιότητα και με την καλύτερη νομοθεσία, το Better Regulation, βλέπουμε πώς εκπονείται η νομοθεσία, πώς εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη και πώς αξιολογείται. Και ενδέχεται να ακολουθήσει σε αναθεώρηση της νομοθεσίας. Υπάρχει το REFIT, που δεν αφορά την απορρίθμιση ή την υποβάθμιση προτύπων, Αντιθέτω, όπως πολύ σωστά είπε η έχει να κάνει με τον έλεγχο, ε, το κατά πόσον εξακολουθεί να είναι επαρκή η νομοθεσία. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την νομοθεσία που έχει να κάνει με το περιβάλλον, μιλάμε για άλλωστε για μεγάλο και εκτιμένο όγκο μεγάλων νομοθετημάτων που πρέπει να εφαρμόζονται σωστά. Πρώτα βλέπουμε αν λειτουργεί λοιπόν και μετά κάνουμε πολύ καλή αξιολόγηση και καταλήγουμε στα συμπέρασματά μας. Στο τη διαφάνεια από δύο λόγια. Γιατί είναι ιδιαίτερα προσφυλέ για σας το θέμα αυτό και ιδίω για τι ΜΚΟ. Φυσικά και έχουμε ήδη πριν από 13 χρόνια θεσπίσει ένα πλαίσιο για την επικοινωνία μας με τους καταγγέλλοντες, τους ενημερώνουμε για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ενημερώνουμε πρωτού λάβουμε για την επόμενη μας απόφαση, δηλαδή όταν κλείνουμε μια καταγγελία, εξηγούμε γιατί και ο καταγγέλων έχει στη τέσσερι εβδομάδε για να αντιδράσει. Και μόνο μετά την παρέλυση αυτή τη προθεσμία κλείνουμε την υπόθεση. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα κεκλεισμένο των θυρών. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει ενημέρωση και μάλιστα μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υπάρχουν οι διοικητικέ εγγύησει. Υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Και βέβαια ενδέχεται αν είναι μια υπόθεση πολύπλοκη και αν έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία με τον ε, καταγγέλλοντα και το κράτος μέλος να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία. Καλό να υπάρχει ένας διαδρόμενος διάλογος με τα κράτη-μέλη. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν βέβαια κάποια στοιχεία, κάποια σημεία αναφοράς και κριτήρια που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε γρήγορα λύσεις. Και αν το κράτος μέλος, το εκάστοτε, δεν εφαρμόζει νομοθεσία, περνάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η κίνηση διαδικασιών επί παραβάση. Στο πακέτο λοιπόν για την καλύτερη νομοθεσία, οι διαδικασίες ε, επί παραβάση είναι μόνο ένα μέτρο, μία οδός. Υπάρχουν και άλλες οδοί, έχουμε θεσπίσει κάποια εργαλεία όπως το ότι επιμένουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βρίσκουν τον τρόπο να εφαρμόσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αφήνουμε κάποια περιθώρια και βέβαια εμεί παρέχουμε συμβουλέ για τη σωστή ερμηνεία τη νομοθεσία. Είναι κάτι που ανέφερε και μια βουλευτή. Η δε προσφυγή στο δικαστήριο δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μέσο ένα από τα μέσα και υπάρχουν και άλλα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το πλαίσιο του πακέτου για την καλύτερη νομοθεσία. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε εμείς, λέει ο Πρόεδρος, και πριν δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτριά μας, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για όσα μόλις είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι θα συζητήσουμε και αυτό το πακέτο, την καλύτερη νομοθεσία, αλλά και το λιγότερη νομοθεσία στο μέλλον που είναι και στο πρόγραμμα της Κομισιόν είναι σαφές ότι θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε την Κομισιόν πώς σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια νέα νομοθετήματα. Ίσως στην προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο. Να ζητάμε όλο και περισσότερο χρόνο ε, να μας αφιερώνει η Κομισιόν, να έρχεται εδώ δηλαδή, για να μας ενημερώνει για το πώς σκοπεύει να εφαρμόζει την νοσιακή νομοθεσία. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν με το σημείο αυτό τη μερικής διάταξη, ξαναδίνω το λόγο στην εισηγήτρια. όπω θέλει να προσθέσει κάτι, κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή και τη συζήτηση, η οποία πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και τα σχόλιά σας χρησιμότατα. Σημειώνω ότι φαίνεται να υπάρχει κοινός παρονομαστής, δηλαδή υπάρχει θέληση να καταπιαστούμε με το πρόβλημα στον τομέα της υγείας και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι σημαντικό εμείς σε αυτή την Επιτροπή να το πιστέψουμε ότι όταν ε, παίρνουμε μια απόφαση μετά από σκληρή δουλειά μαζί με τους πολίτες στη χώρα του ο καθένας, ότι αυτή η νομοθεσία θα ισχύει και ότι η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο θα είναι αποτελεσματικό. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνείτε. Για τις τροπολογίες Χαίρομαι που μου λέτε ε, πώς θα κινηθείτε ως ΕΛΚ για παράδειγμα. Κατάλαβα δηλαδή τη γραμμή πλεύση σας. Θα προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη, να δούμε σε ποιο βαθμό θα συμπορευθούμε. Παράλληλα υπογραμμίζω την σημασία αυτών που έχω καταγράψει ήδη στη γνωμοδότηση. Το θέμα της αύξησης του ρήφητη για την απλούστευση κανόνων ε, συνεχίζεται αυτό το gold plating υπάρχει πολύ μεγάλη ε, φιλοδοξία στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Μην μπερδεύουμε τις βελτιώσεις, ε, η απλούστευση ε, για παράδειγμα είναι ένα πράγμα και κάτι άλλο το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση φιλοδοξιών για το περιβάλλον και την υγεία είναι άλλο. Γιατί αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων και των περιβάλλων. Αυτά είναι τα βασικά. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να προκύπτει από την γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ για αυτά που μου είπατε και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εδώ 29 Μαΐου είναι η προθεσμία, όχι, μισό λεπτό να το δούμε. Ναι, 19 Μαΐου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Στη ψηφοφορία στην Επιτροπή Ένβη στις 15 μέχρι 17 Ιουνίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Κιούρη τον Ιούλιο. Και μετά θα πάει στην Ολομέλεια. Και τώρα, επόμενο και τελευταίο σημείο στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106. Αφαίρεση από τον κατάλογο της Ένωσης ορισμένων αρωματικών ουσιών. Την ένσταση υποβάλλουν οι συνάδελφοι Ρενάτε Ζόμερ και Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη. Η Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη θα λάβει το λόγο για να εξηγήσει τους λόγους της ένστασης. Ευχαριστώ. Προφανώς μιλώ και ονόματι της συναδέλφου Ρενάτε Ζόμερ που δεν μπορεί να παραστεί. Εξεργάζεται άλλα θέματα. Νομίζω συνεδρία σκιωδών και δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας αλλά είμαι εδώ να στηρίξω αυτή την ε, ένσταση. Ε, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αφαιρέσει πέντε σημαντικές αρωματικές ουσίες από τον κατάλογο των ουσιών που έχουν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέντε ουσίες αφορά που χρησιμοποιούμε σε πάνω από 2.000 και ε, αρώματα και αφορά 16 διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και είναι σημαντικό αυτό, νομίζω ότι χρειαζόταν να το υπεθυμίσουμε ότι αυτή η απόφαση δεν είναι αιτιολογημένη καθόλου. Δεν αναφέρεται ο ελάχιστος κίνδυνος που συνδέεται και αφορά την υγεία. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αιτιολόγησή της λέει ότι η απόφασή της δεν έχει καμία σχέση με, καμία, με κανένα κίνδυνο που αφορά τη δημόσια υγεία και εξαρτάται απόλυτα από κάποιες τεχνικής φύσεως θέματα και δικαστικά θέματα. Αυτές οι πέντε ουσίες, οι αρωματικές, είναι από τη δεκαετία του στην αγορά και θεωρούνται ασφαλείς και από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και από άλλους επιφανείς φορείς αξιολόγησης μεταξύ των οποίων παραθέτω την Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Παγκοσμίου Οργάνωσης ε, Υγείας και της οργάνωσης το ΙΕ για την διατροφή και τη γεωργία. Πέραν αυτού υπάρχει και μια άλλη πτυχή που κατά την ε, άποψή μας ε, στηρίζει την ένστασή μας, αυτό που συνδέεται με την αρχή της αναλογικότητας και η δέσμευση για καλύτερη νομοθεσία που τα αναφέρατε πριν πρόεδρε στο προηγούμενο σημείο είναι προφανές ότι έχουμε καθήκον να εγγυηθούμε τα πρότυπα και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ισχύουν, όμως πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τις πέντε ουσίες αυτές, έχουμε μόνο το γεγονός ότι οι προθεσμίες προβλέπονται από τη διαδικασία δεν έγιναν σεβαστές. Στο δεύτερο βήμα αν θεωρήσουμε ότι είναι μόνο πέντε αυτές οι ουσίες που δεν έγιναν διαδικασίες εγκαίρως, πέντε από τις 2.500 2.500 ουσίες για τις οποίες η βιομηχανία, ο τομέας έδωσε εγκαίρως τα στοιχεία, βλέπουμε ότι ο τομέας αυτός ε, κινήθηκε σωστά, έγινε κάποιο τόπιμο σε αυτήν την περίπτωση. Εμεί δεν περιοριζόμαστε μόνο στον έλεγχο των εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όταν χρειάζεται να υπενθυμίζουμε και την αρχή τη αναλογικότητα. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να το θίξουμε αυτό, διότι κατά την άποψή μας θα αντιμετωπίζαμε μια υπερβολική εφαρμογή ή πάρα πολύ αυστηρή της νομοθεσίας που ισχύει θα έχουμε μόνο ζημία στους εργαζομένους και στη βιομηχανία χωρίς να έχουμε κανένα όφελος για τους ε, καταναλωτές. Θα ήταν πολύ επιζήμιο να απαγορευτούν οι πέντε αυτές ουσίες και θα είχα μια βιομηχανία που θα επιβαρυνθεί από κόστος ή υποχρέωση αναδιοργάνωσης. Ε, γνωρίζουμε ότι η αρωματοπία απαρτίζεται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ίδιο ισχύει για όλο τον τομέα των τροφίμων, όπου εκεί βλέπουμε χιλιάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων να υπάρχουν. Λαμβάνοντας υπόψη το ύψιστο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας του τομέα των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύω ότι η αρχή του better regulation θα πρέπει να το διαφυλάξουμε για να εγγυηθούμε σε επιχειρήσεις μας τη συνέχιση της ανταγωνιστικότητάς τους και ίσως και ελπίζουμε να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις εργασίας, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Θα θέλαμε να ζητήσουμε δοθέντως ότι τα στοιχεία που ζητήθηκαν δόθηκαν στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και είναι αναμονή να πάνε στην ΕΦΣΑ για να γίνουν οι αναλύσεις. Ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την πρόταση κανονισμού της πριν να συνεχίσει βάση μιας αποφάσεως που θα είχε συνέπειες αρνητικές. Το επαναλαμβάνω αυτό. Πιστεύω πραγματικά ότι στο πλαίσιο της έφτραυστης πολυέθεσης ανάκαμψης θα ήταν σωστό να το αναφέρουμε αυτό και θα ήταν και ο καλύτερος, ο πιο φυσικός δρόμος να ακολουθηθεί για τη στατηγική που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από παλιά υποστηρίζει. Δηλαδή θέλει να θεωρήσει την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας ότι είναι θέματα που έχουν ύψιστη προτεραιότητα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μέλιορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πέντε είναι οι αρωματικές αυτές ουσίες, ε, η φύση τους είναι η ίδια, χημικά παρασκευάζονται, αλλά η προθεσμία δεν ξεπέρασε κανένα δύο μήνες μόνο από τη βιομηχανία, αλλά πάνω από ένα χρόνο καθυστέρησαν. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε δίκιο αυτό είναι ένα γραφειοκρατικό τεχνικό επιχείρημα. Και αφορά αυτό που λέμε ότι πρέπει να νομοθετούμε καλύτερα. Όμως με ενδιαφέρει κάτι άλλο, όχι το γραφειοκρατικό τεχνικό κομμάτι. Εμένα κυρίως με ενδιαφέρει αυτό ο φόβος που εκφράζεται σε σχέση με τη χρήση αυτών των πέντε ουσιών, γιατί λέει ότι έχει ε, γενοτοξική επίδραση. Οπότε εδώ μπαίνει θέμα υγείας των καταναλωτών. Και η εταιρεία που τα φτιάχνει λέει ότι αυτές οι ουσίες και χρησιμοποιούνται πάνω από 40 χρόνια καμιά φορά στην αγορά και ο ΠΟΗ και ο ΦΑΟ ε, τις κατατάσσει ε, ε, τρεις από τις πέντε για τις οποίες μιλάμε μπορεί ενδεχομένως όμως να έχουν και το φοβάται αυτό η Κομισιόν να έχει γενοτοξικές επιπτώσεις ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων ε, ανέθεσε να γίνουν και άλλες μελέτες και η Κομισιόν λέει ότι ο ΠΟΗ και ο ΦΑΟ αυτές τις επιφυλάξεις για τη γενοτοξική δράση τις συμμερίζονται. Ας μας βοηθήσει λοιπόν η Κομισιόν για τα περαιτέρω, γιατί δεν θα ήθελα να συμφωνήσω εύκολα αν δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η κακή τοξική επίδραση και ποια είναι η θέση της ΕΦΣΑ. Have you something to say? Έχετε κάτι να πείτε εσείς. Ναι, κοιτάξτε, η πρότασή μου ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα να μιλήσει, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις, λέει ο Μπράντι, και ίσως οι περισσότερες θα μπορούσαν να απαντηθούν από την Κομισιόν και να μην καταθέσουμε όλοι τις ίδιες ερωτήσεις, γιατί εγώ τουλάχιστον θέλω κάποια διευκρίνηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση, για παράδειγμα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρόεδρος. Όταν προβάλλουμε μια ένσταση κάπου, ακούμε συνήθως πρώτα τους βουλευτές και μετά παίρνει το λόγο η Κομισιόν. Βέβαια, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, ίσως μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πρώτα σε αυτά που είναι οι δύο συνάδελφοι και να αντιδράσουμε εμείς εν συνεχεία και να κάνουμε τα περαιτέρω τυχόν σχόλια που έχουμε. φωνή λοιπόν, λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέστρατη για κάπω έτσι που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μάλιστα είναι ε, μονάδα, και θα μπορούσε στη συνάδελφο Γκαρντίνα και Μιλιόρ να δώσει κάποιες απαντήσεις και εμείς να μιλήσουμε μετά και να θέσουμε δεχομένως πρόσθετα ερωτήματα αφού θα έχουμε ακούσει τι έχει να μας πει η Κομισιόν αρχικά. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όπως ε, είπαν ε, οι προλαλήσασες, ίσως καλό είναι να δώσουμε το ιστορικό αυτού του σχεδίου κανονισμού που ε, αποσύρει πέντε αρωματικές ουσίες από, την, από τον κατάλογο. Λοιπόν, αυτός ο κατάλογος ήδη από το 2000 ε, είχε υπο, υπαρθεί σε μία αξιολόγηση ανά πέντε χρόνια. Έχουμε ένα κανονισμό το 96 και έχουμε και τον κανονισμό 3034 το 2008 για τις αρωματικές ουσίες και ρύθμιση από το Ευρωπαϊκό, ο κανονισμός μάλλον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τροποποιεί την προθεσμία για την κατάρρευση του νοσιακού καταλόγου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2010 Πριν είχαμε ένα μητρό αρωματικών νησιών μόνο. Αυτός ο νησιακός κατάλογος αρωματικών νησιών ε, λοιπόν θεσπίζεται με τον κανονισμό 872 του 12 της Επιτροπής και περιλαμβάνει περίπου 2.500 αρωματικές ουσίες μεταξύ των οποίων θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθούν 411 ουσίες για τις οποίες ε, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η εξολόγηση κινδύνων και για τις οποίες ζητούνταν ή απαιτούνταν περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία, ορίζονταν οι προθεσμίες στον κανονισμό, εντός ε, των οποίων θα έπρεπε να έχει γίνει αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ και για τις οποίες χρειάζονταν πληροφορίες για να μπορεί να κάνει η ΕΦΣΑ την ε, αξιολόγηση αυτή και στον ε, κανονισμό ξεκάθαρα αναφερόταν ότι αυτό είναι προϋπόθεση, δηλαδή πρέπει να έχει δοθεί η απαραίτητη ενημέρωση μέχρι την λήξη της προθεσμίας και αν δεν είχε δοθεί μέχρι τότε η απαραίτητη ενημέρωση, οι αρωματικές ουσίες εν λόγω θα έπρεπε να αποσυρθούν από τον νοσιακό αυτό κατάλογο. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, γιατί αναφέρθηκε ε, ότι είναι ένα αμυγός γραφειοκρατικό μέτρο, δεν θα το έλεγα έτσι εγώ διότι σε ό,τι αφορά τι αρωματικέ αυτές ουσίες η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή την Ασφάλεια των Ορφών, είχε κάποια ερωτηματικά ως προς την ασφάλειά τους. Γι' αυτό και ήδη από το 2011 είχαν ε, τεθεί κάποιες προϋποθέσεις γιατί χρειαζόταν να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες. Και όπως είπα είχαμε διάφορε προθεσμίε και για αυτέ τι πέντε ουσίε που εξετάζουμε επί του παρόντος είχαμε ε, θεσπίσει την ε, αργότερη δυνατή προθεσμία 31 Δεκεμβρίου 2013 συγκεκριμένα. Μέχρι λοιπόν 31 Δεκεμβρίου 2013 για τις πέντε αυτές αρωματικές ουσίες δεν λάβαμε καμία ε, νέα μελέτη επιστημονική από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τροφίμων. Βέβαια, μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβλήθηκαν εκθέσεις, όπως τον Νοέμβριο ή τον Ιανουάριο ε, του τρέχοντος. Για μία μάλιστα από αυτές τις δεν έχει υποβληθεί ακόμη καμία μελέτη. Όμως προβλέπει ο κανονισμός ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας νέες αιτήσει μπορούν να υποβληθούν δυνάμει του τρέχοντος συστήματος γιατί αλλάζει το σύστημα από το 2010. Έχουμε την κοινή διαδικασία διοδότης πλέον. Όπως είπα λοιπόν, για μια από τις ουσίες δεν έχει υποβληθεί καμία μελέτη, όπως είπα, για τις άλλες έχουν υποβληθεί μελέτες. Αλλά ένα χρόνο μετά την παρέλευση προθεσμίας. Είπα επίσης ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσαμε τη διαδικασία απόσυρσης των ουσιών αφού πρώτα ενημερώσαμε και συγκεκριμένα το Μάρτιο 2014 τους διάφορους φορείς και πρωτοσυζητήσαμε το μέτρο με τα κράτη-μέλη, τις ομάδες εργασίας. Όταν οριστικοποιήθηκε αυτό, η πρόταση, δηλαδή το σχέδιο πρότασης, ε, το υποβάλαμε και στο SPS. Γιατί έχουμε την ε, συμφωνία αυτή για τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά Έπειτα υποβάλαμε στον ε, ΠΟΗ, στον ΠΟΕ συγγνώμη, τα σχετικά και είδαμε και το θέμα της ενδεχόμενης τρέβλωσης της αγοράς ή διαταραχής αγοράς και γι' αυτό προβλέψαμε για τις πέντε αυτές ουσίες μια εννιάμινη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή ακόμη και αφού εγκρίθηκε αυτό το μέτρο, τρόφιμο περίχαν αυτές τις αρωματικές ουσίες θα μπορούσαν να παραμείνουν στην αγορά ή μπορούν να διδεθούν στο εμπόριο μέχρι και εννέα μήνες μετά τη θέση ισχύ αυτού του μέτρου. Άρα έχουν τη δυνατότητα οι παρασκευαστές, ε, παραγωγή αυτών των τροφίμων να ε, προσαρμοστούν. Τώρα, τα επιστημονικά στοιχεία ε, δεν είναι απλά γραφειοκρατικά και τα έχουμε διότι πραγματικά υπάρχουν ανησυχίες όπως την ασφάλεια. Και αν θέλουμε πράγματι να διατηρήσουμε ψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών, δεν θα πρέπει αυτό να το επιδεινώσουμε επειδή είναι απρόθυμοι οι φορείς να μας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Και μάλιστα εγκαίρως, όπως είπα λοιπόν, και οι μελέτες αυτές πλέον έχουν υποβληθεί. Δεν είναι βέβαιο όμως σε ποιο βαθμό θα άρουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια που έχουμε για αυτές τις ουσίες. Που όπως είπα ΕΦΣΑ δεν τις έχει ακόμα αξιολογήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναλογικό το μέσο αυτό διότι και ο κλάδος, ε, οι φορείς θα μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα να αποφύγουν ε, την ε, διαταραχή στην αγορά αν είχαν δώσει τα στοιχεία εγκαίρως, κάτι που δεν έπραξαν, ή να υποβάλουν ήδη τη νέα αίτηση υπό τη νέα διαδικασία της κοινή αδειοδότησης. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό πριν από πέντε μήνες, αφού έχουμε στη διάθεσή μας τις μελέτες. Ούτε και αυτό το έπραξαν όμως. Ένα άλλο σημείο είναι ότι πρέπει να δούμε ότι είχαμε 411 ουσίες στο 11 που υπάγονταν ακριβώς στην ίδια ε, περίπτωση. Δηλαδή έπρεπε για αυτές να υποβληθούν ε, πρόσθετες μελέτες. Υποβλήθηκαν για τις 406 από αυτές και όχι για τις 5. Άρα για 406 αρωματικές ουσίες, οι σχετικοί κλάδοι, οι σχετικές κατέβαλαν την προσπάθεια να δώσουν ε, τα στοιχεία, να διενεργηθούν οι απαραίτητες μελέτες. Άρα δεν ε, προβλέπεται τουλάχιστον στο παρόν στάδιο απόσυρση των εν λόγω ουσιών και θα συνιστούσε άλλωστε αυτό διακριτική μεταχείριση κατά ε, των ε, βιομηχανών που έκανε τις προσπάθειες και υπέρ αυτών που δεν έκαναν αυτή την προσπάθεια και θέλουν τα προϊόντα τους να διατηρηθούν στην αγορά. Ενώ οι άλλοι κλάδοι έκαναν τις προσπάθειες και έδωσαν τα απαραίτητα τι τις μελέτες που έλειπαν. Το μέτρο λοιπόν θεωρούμε ότι έχει απλά ένα αναλογικό, δεν είναι και διακριτικό. Είναι δίκαιο. Αυτά. Ευχαριστώ. Okay. Ε... Καλώς. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Ικανοποιούμε από την απάντηση της Κομισιόν. Αν αυτό σημαίνει η καλύτερη νομοθεσία ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται τίποτα και αν ε, η βιομηχανία μπορεί να κρύβεται πίσω από τις μικρομεσαίες ότι θα είναι πάντα ασφαλής και αν λένε ότι ε, ήταν χρόνια στην αγορά και το DDT ήταν χρόνια στην αγορά για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Εγώ πολύ το εκτιμώ ότι η Κομισιόν παίρνει στα σοβαρά την ε, ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό το better regulation συχνά το μεταφράζει όμως no ή less regulation. Αλλά χαίρομαι που πιστεύετε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να νομοθετούν καλά, καλύτερα. Και αυτό γίνεται με πολύ φιλελεύθερο τρόπο. Αν οι βιομηχανίες θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, θα μπορούσαν να τα έχουν ετοιμάσει όλα αυτά. Και κάτι που με ενόχλησε όταν πρωτοεκλέχτηκα στο Κοινοβούλιο με, πριν από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια ε, στο Εθνικό, είναι ότι ο, ο χρόνος δεν λαμβάνει την υπόψη σωστά. Συσσωρεύονται οι καθυστερήσεις, όλοι καθυστερούν να έρθουν και όλα αυτά ε, στο τέλος έχουν ένα σωρευτικό αποτέλεσμα. Όχι εσείς, απευθυνόμενοι στον πρόεδρο, πάντα είστε στην ώρα σας. Αλλά πολύ συχνά συμβαίνει. Και άμα λέμε, δεν «Ναι, μας νοιάζει η ώρα, δεν πειράζει, θα, τα, θα συνεχίσουμε έτσι. Εγώ πολύ εκτιμώ ότι υπευλήθη η πρόταση αυτή, γιατί όλα αυτά τα ξεκαθαρίζει, ότι οι δουλειές πρέπει να γίνονται σωστά. Δεν θα μπω στην ουσία, ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια, από ό,τι βλέπω υπάρχουν κάποια κίνδυνη. Αλλά μιλάω γενικά, θα πρέπει να μην κρυβόμαστε ε, πίσω από κάποια ε, στοιχεία που ίσχυαν μέχρι τώρα. Πολλές φορές βγαίνει μπροστά μια μικρομεσαία επιχείρηση και αν το ξύσουμε λίγο βλέπουμε ότι από πίσω κρύβεται μια μεγάλη ε, φαρμακευτική εταιρεία. Πρέπει να τα παρακολουθούμε και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και παραδείγματα καλής νομοθεσίας και όχι μόνο να μιλάμε για την κακή νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Φρέντρικ Κρίσ που είναι ο σκιώδης μας και δεν μπόρεσε να έρθει. Ομολογώ ότι το μπαλεύω το φάκελο και δεν έχω καταλήξει, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω κάποια συμπληρωματικά την Κομισιόν. Κατάλαβα, σας κατάλαβα καλά ότι, που είπα, ότι είπατε ότι με αυτές τις πέντε ουσίες υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια και γι' αυτό δεν θα επιτρέπονται πια στην αγορά. Αν ναι, υπάρχει και μια μεταβατική περίοδος ε, του ενός μήνα που φαίνεται 9 μήνες που φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητική. Εξηγήστε μας λίγο καλύτερα λοιπόν τους κινδύνους και γιατί είναι αρκετά μεγάλη αυτή η κίνδυνη θεωρείται ώστε να μην επιτρέπονται στο μέλλον να κυκλοφορούν στην αγορά οι ουσίες ενώ είναι ασφαλές να παραμείνουν για το επόμενο εννιά μήνους στην αγορά. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ε, δεύτερον, υπήρχε κάποιος χρόνος, η προθεσμία ήταν το Δεκέμβρη του 2013, υπήρχε χρόνος λοιπόν οι κατασκευαστές αυτών των ουσιών να υποβάλουν τις απαραίτητες μελέτες και πληροφορίες. Γιατί δεν το έπραξαν Μιλάμε για πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν, δεν γνώριζαν κλπ. Ίσως και αυτό πρέπει να το δούμε. Η τελική μου ερώτηση, η τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι αυτά συζητήθηκαν στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο συμφώνησε να μην επιτρέψει πια να κυκλοφορούν οι ουσίες στην αγορά. Έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο, ψηφίσανε εκεί στο Συμβούλιο ή ελήφθη ομόφωνα απόφαση να ε, συμφωνήσουν με την πρόταση της Κομισιόν εδώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ακούγοντας τις εξηγήσεις των διαφόρων, ε, η ασάφεια επικρατεί. Εκπλήσωμαι κάπως. Δεν συμμερίζομαι την άποψη κάποιων συναδέλφων. Και αυτό διότι οι πληροφορίες που διαθέτω δείχνουν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν ήταν σε θέση να δώσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εγκαίρως. Αντίθετα από αυτό που είπαν κάποιοι, πρέπει να ξέρουμε ότι στη Νότια Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα των αρωμάτων και των διαφόρων αρωματικών ουσιών για τρόφιμα και δεν ανήκουν σε μεγάλους ομίλους. Μην το φαντάζεστε αυτό. Θα μπορούσε να αποφευθεί το πρόβλημα διότι είναι πιο ισχυρές εταιρείε αυτές από ό,τι νομίζετε. Είναι σφαλμένο στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Υπάρχουν πολύ μικρέ μικρομεσαίες επιχειρήσει που κινούνται σε αυτό το τομέα. Θέτω ερωτηματικά μας είπατε ότι υπάρχει μία ουσία για την οποία δεν υπευλήθη κάποια μελέτη, για άλλες ε, υπευλήθησαν εκθέσεις και μελέτες ε, καθυστερημένα και η ΕΦΣΑ από ό,τι κατάλαβα δεν γνωμοδότησε ακόμα. Εν τη αυτή περιπτώση ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε να έχουμε τις πληροφορίες. Πριν πάρουμε ξαφνικά μια απόφαση απόφαση οικονομικής φύσεως που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύο προβλήματα διαβλέπω. Πρώτα απ' όλα, είτε έχουμε μια καθυστέρηση που μπορεί να εξηγηθεί, εν τη αυτή περιπτώσει, στη λογική της καλύτερης νομοθεσίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Διότι στο Κοινοβούλιο επί σειρά ετών ακούω να λέει ο κόσμος ότι πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουμε κλπ. Και όταν προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε κανείς δεν τις στηρίζει ή ελάχιστη. Είτε λοιπόν είναι ένα πρόβλημα καθυστέρησης, σας περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΦΣΑ. Αν η ΕΦΣΑ πει ότι μετά από μελέτε, σοβαρές μελέτες, κάποια αρωματική ουσία για τα τρόφιμα δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας, τότε επανεξετάζουμε το πρόβλημα. Σήμερα όμως δεν έχουμε καθόλου τέτοια στοιχεία. Εγώ στηρίζω στοιχεία που έχουμε. Καλύτερο είναι να περιμένουμε και να μην επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις. Στηρίζω τους συναδέλφους μου και τη συνάδελφο Γκαρντίνη που τοποθετήθηκε πριν. Έχω αμφιβολίες με πληροφορίες που μας έρχονται και είναι αντιφατικές χωρίς διαφάνεια, πώς να τοποθετηθούμε. Από πλευρά τη βιομηχανία, των μικρομεσών επιχειρήσεων έχουμε εντελώ διαφορετικέ πληροφορίε. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε μία γνώμη, την πιο δίκαιη, την πιο ισορροπημένη, την πιο αντικειμενική. Και αυτό που θέλω είναι και ζητώ να υπάρξει περιθώριο προβληματισμού πριν ληφθεί η αδίποτε απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντελαχάη. Η ε, κυρία Τλαχάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να μακρηγορήσουμε. Τα είπε η Φρανσουάς Γκροστέτε, της ουσίας, αυτά που είχα να πω. Απλά ευχαριστώ την προσοχή των συναδέλφων στην ακόμα αρνητική εικόνα που μπορούμε να στείλουμε στους οικονομικούς παράγοντες και στους συμπολίτες μας αν δεν μπορούμε να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Η ΕΦΣΑ θα πρέπει να μας πει ότι οι πέντε αυτές ε, ουσίες είναι επιβλαβείς ή αν δεν είναι επιτέλους πια. Ας ε, πάψουμε με αυτή την γραφειοκρατική διοικητική ακαμψία. Αν και εντάξει, κατάλαβα ε, τι μας είπε η Κομισιόν που αυτός είναι και ο ρόλος της τελικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Στη διάρκεια της συζήτησης λάβαμε και άλλες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον εκπροσωπό της για να τις απαντήσει και αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να τονίσω ότι οι προθεσμίες για την υποβολή των μελετών οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό 872 του 2011 παρήλθαν, γι' αυτό προβλέπαμε διαφορετικές προθεσμίες μετά από διαβούλευση με τον κλάδο για να μπορούν και αυτοί να μας δώσουν τελικά τις ε, μελέτες εντός προθεσμίας. Το 2012, στον κατάλογο, παραλαμβάνω, είχαμε 411 ουσίες που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, ή εξακολουθούσαν να είναι υπό αξιολόγηση ή έπρεπε να υποβληθούν μελέτες. Μόνο για τις πέντε αυτές συγκεκριμένες δεν είχε υποβληθεί μελέτη. Δεν σημαίνει δηλαδή ε, ότι ήταν παράλογη απέτηση, γιατί οι 406 άλλες ουσίες δεν ε, αθέτησαν ε, αυτούς τους όρους. Δεν ξέρω αν το είπα καλά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε ακόμη αποδείξεις ή ενδείξεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, δεν έχουμε αποδείξει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά ότι και δεν είναι επικίνδυνες αυτές οι ουσίες, γι' αυτό είναι απαραίτητο να δεξαχθούν αυτές τις πρόσθετες μελέτες και να δούμε μετά την αξιολόγησή τους κατά πόσο αυτές οι αρωματικές ουσίες δημιουργούν κίνδυνο και πρέπει να αποσυρθούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή υποβλήθηκαν μελέτες πρέπει να παραμείνουν. Ή βάσει των μελετών να συναγάγει η ΕΦΣΑ ότι οι ουσίες αυτές τελικά είναι ασφαλείς. Προς το παρόν όμως, όταν λέω υπάρχουν ανησυχίε ασφάλεια, το λέω γιατί δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσον είναι ασφαλεί ουσίε, χωρί να έχουμε ακόμη στοιχεία ότι είναι επικίνδυνε. Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις, γιατί στη μόνιμη επιτροπή το συζητήσαμε, ψηφίστηκε το μέτρο σχεδόν ομόφωνα. Συγκεκριμένα από τα ε, από τα 28 κράτη-μέλη, τα 27 ήταν υπέρ και απήχε ένα μόνο. Και το λέμε και στην ιστοσελίδα μας για λόγους που σχετίζονται με την αναλογικότητα του μέτρου. Αλλά η στρεπτική πλειοψηφία των κρατών μελών υπερψήφισε το μέτρο. Και αφού πρόκειται για ρυθμιστικό μέτρο, ρυθμιστική διαδικασία, Συμβούλιο θα το έχει ως άλφα σημείο την επόμενη εβδομάδα. Και νομίζω θα αποφασίσει ότι δεν θα αντιταχθεί σε αυτόν τον κανονισμό. Όχι, νομίζω δεν θα αντιταχθεί στον κανονισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τη διακριτική μεταχείριση ή μη. Είχαμε αυτές τις μελέτες εμπρόθεσμα για, εμπρόθεσμα, συγγνώμη, για τις 406 άλλες ουσίες Και δεν είναι μόνο θέμα διακριτική μεταχείριση, είναι και θέμα αξιοπιστία Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέμε ότι ε, καταρτίζουμε ένα νοσιακό κατάλογο, υπάρχουν προϊόντα που είναι ασφαλή, ε, εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και στο Συμβούλιο, υπάρχει διαδικασία με τι οποίε κάποια προϊόντα μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν τον κατάλογο και υπάρχει διαδικασία για την απόσυρση ουσιών από τον κατάλογο ή διαδικασία για το κατά πόσον και με ποιες προποθέσει παίρνουν άδεια οι ουσίες αυτές εγκρίνονται. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με τη βιομηχανία τους ενημερώσαμε ότι είχε λήξει προθεσμία και ότι οι μελέτες δεν είχαν υποβληθεί και το σχόλιο ήταν «Α, δεν είχαμε φανταστεί ότι παίρνει τόσο σοβαρά τις προθεσμίες της Κομισιόν, μα ξέρετε, είναι σε κοινοτική νομοθεσία οι προθεσμίες αυτές». Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό να τι παίρνουμε στα σοβαρά. Και παραλαμβάνω λοιπόν και θέμα αξιοπιστία. Έχουμε καταρτήσει ένα σύστημα, ήταν επαρκέστατε οι μεταβατικές περίοδοι, όπως σα είπα είναι από το 2000. Και προβλεπόταν το 2005 ε, να λήξει προθεσμία, αναβλήθηκε με το 2010 και παραλαμβάνω προβλέπαμε μεταβατική περίοδο για 411 ουσίες, περιμέναμε να υποβληθούν μελέτες. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν, να τελειώσουν αυτές οι περίοδοι μετάβασης. Ήμασταν αρκετά ευέλικτοι μέχρι τώρα, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία του συστήματος. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι okay, δεν πληρούνται προϋποθέσεις, από μέσα αυτά τα περίοδο θα πρέπει να αποσυρθούν από τον ενωσιακό κατάλογο. Δεν σημαίνει απόσυρση όμως ε, ότι γίνεται αυτό για πάντα. Πάντα μπορεί ο κλάδο να υποβάλει μια νέα αίτηση. Έχει τη δυνατότητα. Θα αξιολογηθεί από την ΕΦΣΑ και αν θεωρηθεί ότι είναι ασφαλές το προϊόν, είναι ασφαλή η ουσία, επανεγκρίνεται και ξαναμπαίνει στον νοσιακό κατάλογο. Ήδη μπορούσαν αυτό να το είχαν κάνει εδώ και μήνε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί καμιά νέα αίτηση. Γιατί να μην περιμένουμε, λέτε, μέχρι να έχει αξιολογήσει τι μελέτε η ΕΦΣΑ. Ακούστε, είναι σαφή η διαδικασία μόνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 μπορούσαν να είχαν υποβληθεί μελέτες αυτές και αξιολογηθεί. Να με τις ισχύουσας τότε διαδικασίας ε, έγκρισης για διοδότηση. Από το 2012 και μετά ισχύει μια νέα διαδικασία διοδότηση, κοινή διαδικασία όπως είπα. Θεσπίζεται με τον κανονισμό 3031 του 2008. Και θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι νέοι κανόνες για την υποβολή αιτήσεων και για την εξολόγηση από την ΕΦΣΑ. Άρα δεν σημαίνει ότι τώρα... Μπορείτε να πείτε ναι, έχει περάσει ένα χρόνο μετά την προθεσμία και αυτέ τι ουσίε μπορούμε να εφαρμόσουμε ακόμη το παλιό σύστημα για να εξετάσει η ΕΦΣΑ αυτού τους φακέλους. Αυτό όμω αντιβαίνει στην όνειση και νομοθεσία. Αν θέλουμε το σύστημα αδειοδότηση να είναι αξιόπιστο και τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο να είναι ασφαλή, και να διατηρήσουμε την καλή εικόνα αυτών πρώτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και όπως είπα αυτό είναι ένα αναλογικό μέτρο γιατί προβλέψαμε ήδη μακρές νομοθετικές περιόδους στο παρελθόν. Όπως είπα ήδη είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση από το 2000 και οι προθεσμίες συμφωνήθηκαν κατόπιν διαβούλευσης με τον κλάδο, με την Ευγανία. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ίσως η Ελιζαμπέτα θα ήθελε να ολοκληρώσει, να προσθέσει κάτι όσον αφορά την ένσταση αυτή. Ευχαριστώ, συντομότατη θα είμαι. Να επαναλάβω λοιπόν. Δεν γνωρίζω αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν είχα τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί τους. Όμως αισθάνομαι ότι προερχόμενοι από μια χώρα που οι μικροσές επιχειρήσεις πολύ συχνά εκπροσωπούνται από πολλές, πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις, ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει μήπως ε, βρισκόμαστε σε μία από αυτές τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μικροεπιχείρηση αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες να προσανατολιστεί μέσα σε μία νομοθεσία που αισθάνεται ότι είναι απόμακρη σε μια γλώσσα εντελώς ξένη και διαφορετικά και είναι εταιρείε που ίσως δεν έχουν ανθρώπινους πόρους που είναι σε θέση να διαβάσουν δύο γραμμές στα αγγλικά ε, ή να προσεγγίσουν μια πραγματικότητα που θα έπρεπε να προσεγγίσουν. Αλλά είναι και αρμοδιότητα της Ευρώπης αυτή να συνοδεύει σε αυτή την αλλαγή που κάποιοι την έκαναν από παλιά, κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές όμως με κόπο προσπαθούν τώρα να ξεκινήσουν να κάνουν την αλλαγή και δεν είναι εύκολο και βλέποντας ότι μόνο πέντε από τις 2.500 ουσίες έμειναν εκτός του χρονικού ορίου ε, δείχνει ότι 99,9% των επιχειρήσεων πέσουν σοβαρά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ίσως όταν έχουμε τόσο μικρό ποσοστό πράγματι να βρισκόμαστε έναντι μιας έλλειψης κατανοήσεως από τις πλευράς των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Κάτι δεν έγινε πλήρως κατανοητό. Τέσσερις από τις πέντε ουσίες, από ό,τι βλέπω, ήδη έχουν μελετηθεί, υπάρχουν μελέτες και θα μπορούσαν ε, να προωθηθούν προς την έψα για να δοθεί μια απάντηση επί της ουσίας. Ίσως μπορούμε να κάνουμε προσπάθεια. Να μπούμε στην ουσία. Να επιβραδύνουμε, να βραχύνουμε το χρόνο ε, της ανάλυσης, προστατεύοντας έτσι και την υγεία των πολιτών που είναι στην πρώτη στη θέση, αλλά και τις επιχειρήσεις. Που δεν είναι τόσο εύκολο να αποσύρουν μια και μετά να την ξαναβάλουν στον κατάλογο. Εάν θεωρούνται από πολλοί μεγάλους διεθνείς φορείς ότι είναι ασφαλείς αυτές τις ουσίες. Ε, μάλλον είναι ουσίες αυτές που δεν δημιουργούν κάποιο κίνδυνο. Υπάρχουν και συνάδελφοι που με στηρίζουν. Ζητώ να εξεταστεί η ουσία του θέματος. Να γίνει μια προσπάθεια. Να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά εμπόδια Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Να υπενθυμίσω. Ψηφοφορία στην Έμβη. 26 Μαΐου. Ολομέλεια. Ιούνιο. Θα υιοθετηθεί το σχέδιο ψηφίσματος. Δεν έχουμε άλλο σημείο στην μισή διάταξη. Ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 στη συνεδρίες Επιτροπής ΕΝΒΗ και στις 9 θα συνεδριάσουν συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο.